ε, θα μιλήσω θα ουγγρικά και θα προεδρεύσω τη συνεδρίαση οπότε επανέρχομαι στην ημερήσια διάταξη σχετικά με τις προφορικές ερωτήσεις που απευθύνονται εις ε, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους. Καλωσορίζω τον Επίτροπο κύριο Κάλλας και τον κύριο Σίμψον, τον συντάκτη της προφορικής ερώτησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ε, ε, σχετικά με την ε, προφορική οδηγία για την εφαρμογή του πακέτου, ξέρετε ότι υπάρχουν τρεις υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες από το 2001 και ε, θα ήθελα τώρα όμως να επανέλθω στο θέμα αυτό με μία προφορική ερώτηση διότι 9 χρόνια μετά συζητάμε διότι 21 κράτη-μέλη μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 δεν έχουν εφαρμόσει αυτές τις ε, οδηγίες. Οπότε ε, νομίζω ότι εφόσον φτάνουμε στην αναθεώρηση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου μία σειρά κρατών τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά ε, και που ε, είναι από τους ενθουσιώδεις προευρωπαδιστές δεν έχουν εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις παρόλες τις διαβεβαιώσεις διαβεβαιώσεις που είχαν δώσει το 2001 στο Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ανησυχητικό και αξιοπερίεργο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουμε να έχουμε μία ενιαία αγορά αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στη, στα θέματα των σιδηροδρόμων και ε, ε, υπάρχουν τμήματα της βιομηχανίας ε, του κλάδου ε, που ενδιαφέρονται αλλά το Κοινοβούλιο πλέον δεν μπορεί να περιμένει διότι υπάρχει ε, η ανησυχία ότι παραβιάζεται εσκεμμένος η νομοθεσία και δεν υπάρχει παρακολούθηση των κρατών μερών. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε ποια κράτη και ποια τμήματα της νομοθεσίας δεν έχουν συμμορφωθεί ε, και ε, τι έχει γίνει. Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία ακόμη ανθίστανται εις την αρχή της, ε, του δίκαιου ανταγωνισμού στον τομέα και εσκεμμένος προσπαθούν να συγκαλύψουν τις ε, ε, εθνικές τους αρμοδιότητες. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες ε, των ανεξαρτήτων διαχειριστών στις χώρες αυτές. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και εναρμόνιση και των χρεώσεων και οδηγεί σε μία προστασία της πρακτικής αυτής και δεν βοηθά στην πρόθεσή της και συγχρόνως ε, ε, καταπιέζει τις ε, δια συνοριακές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε αν ορισμένα από τα κράτη αυτά είχαν ποτέ την πρόθεση να εφαρμόσουν καν αυτές ε, τις οδηγίες και τώρα θα θέλαμε να ξέρουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, πώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αναμόρφωση του κειμένου θα μπορέσει να εφαρμόσει το πακέτο των σιδηροδρόμων. Τι θα κάνει η Επιτροπή για να εφαρμόσει στην την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτό. Θα θέλαμε να ξέρουμε γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να στραφεί η Επιτροπή προς τις ε, χώρες που δεν έχουν συμμορφωθεί. Διότι η Επιτροπή ε, Μεταφορών αναφέρεται πολύ σε την διασύνδεση των σιδηροδρόμων μεταξύ κρατών διότι διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσει να υπάρξουν διευρωπαϊκές συγκοινωνίες επιβατών και η αγορά εμποδίζεται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πραγματική προοπτική ε, του δικτύου και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το πακέτο των συνδυροδρόμων. Εάν δεν ληφθεί αυτό το πρώτο μέτρα, τα επόμενα δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε άμεση δράση και να την έχουμε τώρα θα έπρεπε να αναφερθούμε στα κράτη και να αναλάβουμε τις σωστές ενέργειες τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Επίτροπος, ο κύριος Κάρλας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Και ευχαριστώ την Επιτροπή Μεταφοράς που προκαλεί αυτή τη συζήτηση. που θέλει να προωθήσει το άνοιγμα και τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των σιδηροδρόμων. Η παρακολούθηση ε, του τομέα που ε, δημοσίευσε η Κομισιόν το 2009 δείχνει ότι σε όλους τους τομείς της αγοράς, ε, μετά το άνοιγμα της αγοράς και την υιοθέτηση του πρώτου πακέτου υπάρχουν ε, θετικές, θετικά βήματα. Όμως η οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις ε, στους σιδηροδρόμους και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχασαν 30% των εργασιών τους. Υπάρχουν δομικά προβλήματα στους σιδηρόδρομους σήμερα. Αυτά τα προβλήματα συνδέονται με τα οικονομικά στοιχεία των σιδηροδρόμων και με οικονομικές αδυναμίες εγγενείς. Διάφορα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, δώσει τα επαρκή κονδύλια για την, στους διαχειριστές των υποδομών. Αυτό ε, σημαίνει χαμηλές υποδομές, προβλήματα στους σιδηροδρόμους. Απ' την άλλη υπάρχουν οικονομικοί και τεχνικοί φραγμοί για την είσοδο στην εισαγορά, όπου οι νέοι φορείς, ε, οι νέες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους υπάρχοντες ε, φορείς που έχουν έμεσο έλεγχο στην υποδομή της υδροδρομική. Ε, τα νέα, οι νέες ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν πάντα τις απαραίτητες εξουσίες και την ε, ανεξαρτησία, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν δίκαιες συνθήκες στην αγορά στην αγορά. Ε, εμείς έχουμε μια διτή προσέγγιση, ε, διαδικασίες επί παραβάση για να αντιμετωπίσουμε την ε, εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων και αλλαγή των κανόνων όταν οι κανόνες δεν είναι αρκετά σαφείς ή ακριβείς. Στο πρώτο επίπεδο, οι διαδικασίες επί παραβάση σημαίνουν λεπτομερή ανάλυση της νομικής κατάστασης και στα 25 κράτη-μέλη ε, στους σιδηροδρόμου και οδηγούμαστε σε αιτιολογημένες νομοδοτήσει οι οποίες εστάλησαν το 2009. Τα βασικά προβλήματα είναι καταρχάς ανεπαρκής εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών καθώς και την πρόσβαση έλλειψη ανεξαρτησία των διαχειριστών των υποδομών και ανεπαρκή ανεξαρτησία, πόρη και, και αρμοδιότητες στους αρμόδιους φορείς. Ε, ε, γι' αυτό ακριβώς αναθεωρήσαμε και ε, ανα, ανακοινώσαμε την αναθεώρηση του πακέτου, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε μια συνολική προσέγγιση, ούτω ώστε να υπάρχει μια πραγματική εσωτερική αγορά για τους σιδηροδρόμους, τεχνική εναρμόνιση στους σιδηρόδρομους, σε συνδυασμό με την σιδηροδρομική υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Γκρός θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι αν ο, ο, ο ζωγράφος Μαγκρίτ είχε ζωγραφίσει τις οδηγίες αυτές θα είχε γράψει από κάτω αυτές δεν είναι οδηγίες Όντως για μένα η όλη συζήτηση την οποία διεξάγουμε εδώ και κάμποσο καιρό είναι σχεδόν σουρεαλιστική διότι έχουμε αποφάσεις ε, οι οποίες λήφθηκαν το 2003 που έπρεπε να έχουν ε, ξεκινήσει να εφαρμόζονται το 2006 και το 2010 ρωτάμε γιατί οι 21 χώρες δεν ε, έχουν συμμορφωθεί σε αυτά τα οποία έχουν υπογράψει. Θα έπρεπε να υπάρχει υπάρξουν ε, νέοι ενδιαφερόμενοι στην αγορά αλλά η εικόνα είναι τελείως διαφορετική και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου είτε είμαστε υπέρ είτε κατά της απελευθέρωσης στον τομέα αυτών πρέπει να κάνουμε μια ε, ε, αξιολόγηση αυτής της απελευθέρωσης η οποία καν δεν έχει εφαρμοστεί οι εταιρείε από την άλλη πλευρά και το είδαμε αυτό σε διάφορες χώρες εν ονόματι της απελευθέρωσης έχουν λάβει αποφάσεις οι οποίες πλήττουν το προσωπικό και τα μέτρα παρόλο που δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι οι ιστορικοί χρήστες των σιδηροδρόμων εμποδίζονται ε, όσον αφορά την τεχνική ε, των ε, σιδηροτροχιών, την αλληλεπίδραση και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανείς να ανοίξει την πόρτα ε, αλλά μάλλον να την κλείνει και αυτό συμβαίνει στις περισσότερες αγορές αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι προτάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί είναι ένα πρώτο βήμα. Για μένα πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση της απελευθερώσεως για να μπορέσουμε σύντομα να υποχρεώσουμε να συμμορφωθούν αυτοί αυτοί οι οποίοι δεν το έχουν ακόμη πράξει και θα πρέπει η Επιτροπή να επέμβει και να δράσει. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκρός. Και τώρα ένα λεπτό ο κύριος Ελ Καντράουι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μερίδιο της αγοράς, της σιδηροδρομικής αγοράς, έχει μειωθεί. Ήταν 30% σε σχέση με το σύνολο των μεταφορών το 82 μετά έπεσε στο 13% και, σταθεροποιήθηκε. Η απελευθέρωση λοιπόν δεν λειτουργεί επαρκώς. Η, το άνοιγμα των αγορών δεν είναι επαρκές. Χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για να πετύχουμε την αύξηση του μεριδίου και σε ό,τι αφορά τις υποδομές και σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την πρόσβαση στην αγορά, τη διαλειτουργικότητα. Χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα και μέσα εκτός της απελευθέρωσης. Αν δεν τα δούμε όλα αυτά με συνεκτικό τρόπο, δεν πρόκειται να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μας είπατε ότι σχεδιάζεται αναθεώρηση του πρώτου πακέτου. Πότε θα την έχουμε και ποιοι είναι οι στόχοι αυτή τη αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ελκαντράουι. Και τώρα δύο λεπτά ο κύριος Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολύ χάρηκα όταν στην ακρόαση στην Επιτροπή Μεταφορών είπατε ότι το καλύτερο που μπορούσαμε να επιτύχουμε στην Ευρώπη ήταν η ελεύθερη διακίνηση και η κινητικότητα των πολιτών. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό δεν πρέπει μόνο τα άτομα να μπορούν να μεταφερθούν από το ένα σημείο στο άλλο αλλά και τα εμπορεύματα. Και ήδη το 1992 είχαμε αποφασίσει ε, να υπάρξει ενιαία αγορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρώπη και το 2001 δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τους σιδηροδρόμους. Τώρα όμως είμαστε στο 2010 και είναι ντροπή ότι 21 κράτη ακόμη μπλοκάρουν και δημιουργούν προσκόμματα. Αυτό έχει σχέση με τον προστατευτισμό, έχει ήδη αναφερθεί και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και λυπηρό που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αναφέρθηκαν τα διάφορα συστήματα σιδηροτροχιών, αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα, υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες πιστεύουν να ξεφύγουν ε, και να παραμείνουν στο παλαιό καθεστώς και να ε, προσπαθούν να διαχωρίσουν τις υποδομές από τις παροχές υπηρεσιών. Πιστεύω ότι ο δρόμος αυτός είναι λανθασμένος και πολύ με ενδιαφέρει να ξέρω Οπότε πρόκειται να ξεκινήσετε την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας και θα ήθελα να σας προτρέψω όπως είπαν και οι προλαλήσαντες να είστε αυστηρός με τα κράτη-μέλη γιατί όλοι συμφωνούμε ότι στο πακέτο αυτό πρέπει να ε, υπάρξει τάξη. Είσαστε νέος επίτροπος, δεν φταίτε για τις παραλήψεις των προκατόχων σας άρα μπορείτε κατευθείαν να προχωρήσετε στο θέμα των σιδηροδρόμων και να μπορέσετε με, ε, να προωθήσετε το θέμα αυτό με τους άλλους Ευρωπαίους. Ελπίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί και προσβλέπω σε αυτό που θα κάνετε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Η κυρία Ιζαμπέλ Ντουγάν για δύο λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, εδώ και 15 χρόνια έχουμε αυτό το πρώτο συνδρομικό πακέτο. Την εποχή εκείνη οι στόχοι ήταν να κερδίσουν μερίδια της αγοράς οι ισοδομικές εταιρείε. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Η απελευθέρωση τη της αγοράς ήταν από τα μέσα και δίνει αποτελέσματα όχι πάντα θετικά. Ε, στην πραγματικότητα ε, υπάρχει στασιμότητα στους σιδηροδρόμους ενώ αυξάνει το μερίδιο των οδικών μεταφορών. Ε, την ίδια στιγμή ο αριθμός των επιβατών αυξάνεται και δεν δουλεύει ο ανταγωνισμός. Επίσης μιλήσατε για νέες ε, επιχειρήσεις, αλλά είναι πολύ λίγες αυτές και πολλές από αυτές έχουν απορροφηθεί από τις μεγάλες εταιρείε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το μονοπόλιο των μεγάλων εταιρεών ήταν ο επιζητούμενος στόχος. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, αν δούμε τις διαδικασίες επί παραβάση, αντικειμενικά ε, υπάρχει πρόβλημα, ιδίω ό,τι αφορά την ανεπάρκεια της ε, ανεξαρτησίας των εθνιστικών αρχών και των αρχών προσφυγών και ακόμα και όταν υπάρχει ε, λειτουργική ή θεσμική διαφοροποίηση. Ε, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα, σε κόστος και σε προβλήματα ό,τι αφορά τον εσωτερικό συντονισμό. Ε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να είσαστε προσεκτικός να προχωρήσετε με μια ολιστική προσέγγιση, να κάνετε μια πλήρη αξιολόγηση των προηγούμενων πακέτων, χωρίς να έχετε προηγημένες αποφάσεις, να κάνετε την αξιολόγηση για να δείτε μετά τι θα κάνετε. Ε, να μην είσαστε συγκαταβατικό, να δείτε τι συνθήκες ασφάλειας, τι ασφα... τις συνθήκες ε, ε, εργασίας, την ασφάλεια την ανεπάρκεια ε, εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστου, να τα δείτε όλα αυτά πριν περάσετε σε μεγαλύτερη απελευθέρωση. Θα ήθελα λοιπόν να δω ποιε είναι οι προτεραιότητες όλου αυτού του τομεί, να λάβετε υπόψη κάποια σημεία προόδου, ε, να δούμε κάποια σημεία διαφάνειας ό,τι αφορά το reporting, την εναρμόνιση των, της κατάρτισης, θέματα που αφορούν τη σηματοδότηση, αλλά θέλω να γίνει μια αξιολόγηση συνετή, χωρίς ταμπού, ούτω ώστε να μην προχωρήσουμε πολύ γρήγορα από εδώ και πέρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Ντουγόν. Και τώρα δύο λεπτά, ο κύριος Βλάζακ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι όταν δημιουργήθηκε το γενικευμένο πλαίσιο για την ρύθμιση των σιδηροδρόμων ελπίζαμε ότι θα είναι πιο διάφανο το μελλοντικό σύστημα. Είχαμε την εντύπωση ότι ο ευρωπαϊκός τομέας των σιδηροδρόμων βρισκόταν ε, στην παραμονή μιας νέας εποχής. Αυτό όμως δεν υλοποιήθηκε. Οι 21 κράτη συμπεριλαμβανομένης και της Τσεχίας δεν εφάρμοσαν το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο και ορισμένα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί σχετικά με το άνοιγμα των αγορών των σιδηροδρόμων. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε και στη τσεχική δημοκρατία. Παρόλο που το κράτος έχει κάνει τα πρώτα βήματα για να ανοίξει την αγορά σε τρίτους, δεν υπάρχει πολιτική θέληση και αυτό οφείλεται στους υπευθύνους σε περιφερειακό επίπεδο και οι οποίοι σύναψαν δεκαετής συμφωνίες με τους τσεχικούς σιδηροδρόμους χωρίς διαδικασία προκηρύξης φύσεως μειοδοτικού διαγωνισμού. Έχουν, έχουν κερδίσει λοιπόν ακόμη πέντε χρόνια, έχουν κλείσει την αγορά για την επόμενη 15 ετία και δεν υπάρχει ε, μία εξέλιξη ε, η οποία θα είναι ούτως ή άλλως μοιραία για το μέλλον των σιδηροδρόμων και αυτό σημαίνει ότι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τώρα απειλούν με απεργίες διότι υπάρχουν προβλήματα και οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι στο περιθώριο της οικονομικής ζωής της χώρας και δεν είναι δυνατόν να μειώσει κανείς τις οδικές μεταφορές τις οποίες κατακρίνουν τόσο πολύ οι πράσινοι. Θα ζητούσα λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιηθεί για να απελευθερώσει τον τομέα των σιδηροδρόμων και θα πρέπει να επιβλέπουμε για να συμμορφωθούν και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στην αγορά. Κόλιτσεκ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ με τον κύριο Βλάσακ διότι η δικιά του κυβέρνηση επίσης συμμετείχε σε αυτά τα οποία ο ίδιος κατακρίνει. Και τώρα ε, ε, βλέπουμε ότι το πρώτο αυτό πακέτο ήταν τρεις οδηγίες που έχει επικυρώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που προωθούσαν το άναγμα της αγοράς διαχωρίζοντας ε, την, τις υποδομές των μεταφορών ε, των εμπορευμάτων από των επιβατών και ε, ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι εν μέρη έχουν καλυφθεί οι στόχοι των οδηγιών χωρίς όμως να έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και με τις συνθήκες εργασίας των σιδηροδρομικών υπαλλήλων υπαλλήλων ε, πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε εάν συνάδει το πακέτο αυτό με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί για να εξετάσουμε συγχρόνως και το εάν έχουν ανοίξει οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να υπάρχει ε, μία δυνατότητα δυνατότητα προωθήσεως περιφερειακής όπως συμβαίνει και στη Γερμανία και δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μία μέθοδος η οποία κρατά ε, ε, επαχθεί συνθήκες ε, για τους εργαζόμενους. Νάτρας, δύο λεπτά. Πρόεδρε, στο το, η κυβέρνησή μας έχει εφαρμόσει το πακέτο. Ε, ενδεχομένως επειδή έχουμε παραχωρήσει εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διαχωρισμός των υποδομών από την ε, διαχείριση έχει δημιουργήσει προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ε, επικρατεί χάο στο δίκτυό μα. Δεν είμαι σοσιαλιστή, αλλά αν θέλουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, ε, σίγουρα καλύτερα το δίκτυο να το κατέχει το κράτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε έξι διαφορετικέ ε, επιχειρήσει ε, ανάμεσα στο Μπέρμιχαμ και το Βερολίνο, στην ίδια γραμμή. Όταν αφήνουμε διάφορες εταιρείες να λειτουργούν πάνω στο ίδιο δίκτυο, δεν έχουμε πια τροχαίο υλικό. Ε, γίνεται αστεία η κατάσταση. Ο κύριο Σίμψον που είναι υπεύθυνο είναι μέλος του Εργατικού κόμματο, πρώην σοσιαλιστής. Και εξελέγει από ανθρώπου που πιστεύουν ακόμα ότι σοσιαλισμό και εργατικό κόμμα είναι το ίδιο πράγμα. Και τι ζητάει. Ζητάει ιδιωτικοποίηση. Αλλά πάνω από αυτό το μοντέλο είναι ένα κοινωτικό μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί. Και σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των ίδιων των εκλογέων του, του ίδιου του εκλογικού του ε, σώματος. Είναι πολύ δύσκολο η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει δεκτή, δεδομένου ότι θα εκτροχιάσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νάτρας. Δύο λεπτά. George Bach. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαιρετίζω την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου και την αναμόρφωσή του. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχει γίνει αυτή η επαλήθευση εδώ και καιρό. Αλλά τυχώς η Επιτροπή υποθέτω δεν έχει επαρκές, επαρκείς πληροφορίες από τα κράτη και είναι δύσκολο να αξιολογήσει. Δεν χρειάζεται όμως μόνο να αξιολογήσει, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να ε, ε, επιβλέψει ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται. Πρέπει να μετρήσει κανείς τα αποτελέσματα, διότι τα τελευταία ε, χρόνια είχαμε αρνητικές επιπτώσεις. Έχουμε αποκομίσει τα συμπεράσματα αυτά, η κατάσταση κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, ιδίω σχετικά με την ποιότητα και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει δεσμευτικά ποιοτικά κριτήρια διότι μιλάμε για χαμηλή ποιότητα αλλά δεν πρέπει να μιλά μόνο κανείς για τις ελλείψεις αλλά και για την έλλειψη χρηματοδότησης παρόλη την χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής βλέπουμε όλο και περισσότερη χρηματοδότηση ε, του οδικού συστήματος από ότι του σιδηροδρομικού. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στους σιδηροδρόμους και ε, στο δικό σύστημα. Επίσης επανέρχομαι τώρα στο θέμα τη της μεταφοράς επιβατών διότι ε, βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει μία τεχνική εναρμόνιση διότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές για να μπορέσει να υπάρξει μία ενιαία εφαρμογή των οδηγιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπαχ. Και τώρα η κυρία Σίλβια Αριάννα Τικάου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να είναι μία προτεραιότητα της Ευρώπης ως το 2020 και θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση και εξέλιξη του σιδηροδρομικού δικτύου. Αλλά δεν πρέπει εδώ να αναφερόμαστε μόνο στην ασφάλεια αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών. Όταν λοιπόν μιλάμε για την εφαρμογή του πρώτου σιδηροδρομικού ηλεκτρονικού δικτύου πρέπει να εξετάσουμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι στον ε, τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών ε, ε, έχουν υπάρξει μαζικές απολύσεις οι οποίες είχαν μία αρνητική επίδραση στην εναρμόνιση. Μέχρι το τέλος του παρελθόντος τους 2.700 χιλιόμετρα ε, σιδηροτροχιών προσαρμόστηκαν αλλά χρειάστηκε να υπάρξουν και μεγάλες ε, επενδύσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, θα χρειαστούν όμως και μεγαλύτερες στο μέλλον. Ο κύριος Τσαρνέσκι, παρακαλώ. Κυρίε και κύριε Επίτροπε, Στην Πολωνία λέμε ότι αν κάποιο σου πει ότι είσαι μεθυσμένο, μπορεί να τον αγνοήσει. Αν όμω πέντε σου πούνε ότι είσαι μεθυσμένο, καλύτερα να πέσει να ξαπλώσει λιγάκι. Λοιπόν, αν μια-δύο χώρε μόνο δεν είχαν εφαρμόσει το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο, τότε θα λέγαμε ότι φταίνουν αυτές. Θα λέγαμε να του επιβληθούν κυρώσει κλπ. Αν όμως 20 χώρε δεν έχουν εφαρμόσει το πρώτο σιδηρονομικό πακέτο, τότε ίσω φταίει το πακέτο. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο συνάδελφο από το Ηνωμένο Βασίλειο το επέκρινε. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε γιατί η εφαρμογή του έχει εκτροχιαστεί. Μερικά ατυχήματα μάλιστα τα συζητήσαμε πριν μερικέ ώρες εδώ, στο ημικύκλιο. Και με αυτόν τον τρόπο περνάω στην ασφάλεια. Η ασφάλεια πρέπει να βελτιωθεί. Ο Επίτροπος Κάλλας είπε ότι πολλές χώρες δεν επενδύουν παρακώς στο σιδηροδρομικό τους δίκτυο. Ότι δεν κατασκευάζουν καινούριες υποδομές. Η Πολωνία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτό το φαινόμενο. Ο προπολογισμό για τους σιδηροδρομικές ε, μεταφορές, για το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μια τρύπα Και δεν χρειαζόμαστε συνθήματα απλοποιητικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ενά, 1,5 λεπτό. Ε, πολλοί θρυνούν τις δυσκολίες ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του πρώτου ε, πακέτου. Εγώ χαίρομαι στην χώρα μου και στην περιοχή μου. Ε, συνεργαζόμαστε με τις ε, επιτροπές των χρηστών ε, και με τα συνδικάτα, ούτως ώστε να μην εφαρμοστεί αυτό το πακέτο. Στη Γαλλία ένα από τα διακυβεύματα των περιφερειακών εκλογών είναι το μπλοκάρισμα από τα περιφερειακά συμβούλια σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ε, των σιδηροδρόμων. Δεν θέλουμε να υπάρχουν σιδηρόδρομοι ε, ιδιωτικοί θέλουμε ε, προσπελάσιμους, γρήγορους, ασφαλείς σειροδρόμους. Ε, δεν θέλουμε ε, σειροδρόμους δύο ταχυτήτων. Κάθε μέρα που περνάει δείχνει ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στην υποδομή και στις μεταφορές που επιβάλλουν οι οδηγίες για να επιτραπεί το άνοιγμα στον άγριο ανταγωνισμό είναι μια τεχνική ηλικιότητα που κοστίζει και στον χρήστη και στον φορολογούμενο. Ε, αποδιοργανώνει τις δημόσιες μεταφορές, είναι υπεύθυνη για την ε, επιδίνωση του δικτύου και την ασφάλεια και οι οδηγίες καταστρέφουν και θέσεις απασχόλησης και απλώς εξυπηρετούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρος Πάσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ η αποδοχή των τριών ε, οδηγιών σχετικά με το πακέτο των σιδηροδρόμων ε, σημαίνει μία εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό διότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή και μπορεί να υπάρξουν ε, άνοδοι της τιμής και συγκεκριμένα προβλήματα αλλά είναι προφανές ότι ε, έχουμε καλή υποδομή και καλά οργανωμένες μεταφορές για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις οδικές μεταφορές οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον. Δεν φτάνει όμως να κοιτάμε μόνο το παρελθόν, πρέπει να κοιτάξουμε επίσης και το μέλλον διότι από τρεις πλευρές τα σιδηροδρομικά δίκτυα καταλήγουν στη θάλασσα. Πρέπει όμως να υπάρχει μια καλή διασύνδεση προς Ανατολάς γιατί θα δινόντουσαν νέες δυνατότητες στο σύστημα. Γι' αυτό και ε, ε, αν μπορούσαμε να επεκτείνουμε ε, το, την ταχεία Παρίσι-Βιέννη προς την Πρατισλάβα θα είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα διότι τότε θα δημιουργόντουσαν νέες πολλές δυνατότητες ε, ε, υπάρχουν και δύο μεγάλα αεροδρόμια ή σε τη Βιέννη και την Πρατισλάβα υπάρχει ο Δούναβης για τις ποτάμιες μεταφορές και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μία νέα μέθοδο μεταφορών στην Ευρώπη στο χώρο αυτό θα δινόταν νέα δυναμική και θα είχαμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε ε, θα έπρεπε να σκεφτούμε για νέες επενδύσεις θα υπήρχαν θετικές επιπτώσεις στον τομέα αυτό για να είναι πιο αποτελεσματικές οι σιδηροδρομικές μεταφορές προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης. Ο κ. Καντσάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτή την περίοδο μιλάμε όλος ιδιαιτέρως για τον προγραμματισμό των μεταφορών και θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό και την επόμενη περίοδο. Θεωρώ ότι είναι αποθαρρυντικό το να ξεκινάμε με αυτό το πρώτο ε, πακέτο και με την αναθεώρηση αυτού του πρώτου πακέτου και να διαπιστώνουμε ότι αυτό που συνέβη μέχρι τώρα είναι ανεπαρκές. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία και για να το καταφέρουμε θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο θάρρος. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε τρία ουσιαστικά σημεία κατά την απόψή μου. Το πρώτο νομίζω ότι είναι η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, ε, κάτι που δημιουργεί και ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισμό και προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν διαφανείς κανόνες ε, και σαφείς κανόνες για όλους. Αυτό το ακούσαμε. Το δεύτερο εστιακό σημείο είναι η διαλειτουργικότητα, η διατροπικότητα μεταξύ των κρατών και των διαφόρων μέσων μεταφορών. Και φυσικά το τρίτο σημείο είναι η ασφάλεια. Θα πρέπει η πιστοποίηση της ασφάλειας να είναι προϋπόθεση για την άδεια των επιχειρήσεων. Ε, στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς δεν αρκεί να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, στα κράτη ε, σε ό,τι αφορά την ε, αναποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών αρχών. Θα πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει την επόμενη περίοδο να κάνουμε αυτή την προσπάθεια όταν μιλήσουμε για την βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών, για την αναθεώρηση των δικτύων TEN, την αναθεώρηση των μεταφορών των φορτίων Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να αντιστραφεί μέχρι τούδε πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καντσάν. Και τώρα ένα λεπτό η Ινές Αγιάλα Σέντερ. Η χώρα μου όπως και άλλες 20 δεν έχουν εφαρμόσει δεν έχουν μεταγράψει ε, το πακέτο αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξεκινήσει. Το πρόβλημα μας κυρίως αφορά τα εμπορεύματα. Σε μια περιφερειακή χώρα που χωρίζεται από μια οροσυρά 500 χιλιόμετρων από την υπόλοιπη Ευρώπη, τα Πυρηναία, που ε, μπορεί να περάσει ο σιδηρόδρομος μόνο από τα δύο άκρα της. Ε, έχει επιπρόσθετα προβλήματα εξαιτία του διαφορετικού πλάτου του δυναμικών γραμμών από τη μία και την άλλη μεριά του, των συνόρων. Ποιο λόγο θα είχαμε να έχουμε περισσότερου του ε, ενό παρόχου υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο, πέραν των κυρώσεων που μας απειλούν, χρειαζόμαστε και το καρότο των, της ε, ενοποίησης του συνδρομικού δικτύου στην Ευρώπη. Με αυτό τον... Επίσης θα χρειαζόμασταν ένα κεντρικό τούνελ ναι, διέλευσης των ε, Πυρηναίων, ε, ιδιαίτερα για τα εμπορεύματα. Χρειαζόμαστε άξονες βορρά-νότου και ανατολής δύση στην Ευρώπη για τη μεταφορά των εμπορεύματων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Και τώρα, πριν περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye, Βλέπω ότι ο κύριος Κίψον, Σίμψον συγγνώμη, ζητάει να παρέμβει για να κάνει κάποιες διευκρινήσεις. Με ανέφερε ένας από τους βουλευτές που είναι αντίθετος ε, στην παράταση, ε, στα όσα πρεσβεύει η παράταξή μου. Ο κύριος Νάτρας ε, ανέφερε τον τομπά μου και συνεχεία έφυγε από την α, συνεδρίαση χωρίς να ακούσει τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχετε και στο μυαλό σας την όλη διαδικασία και τον τρόπο που διεξάγεται η διαδικασία. Εγώ παρουσίασα την προφορική ερώτηση εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών ως πρόεδρός της ε, και είναι το καθήκον μου να κάνω κάτι τέτοιο. Υπ' αυτή την έννοια την ε, υπέβαλε. Επομένως δεν νομίζω ότι θα πρέπει η άλλη παράταξη του Κοινοβουλίου να με στυλιτεύει και να με κακομεταχειρίζεται. Πάντως, το... τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ισοδομικές μεταφορές και στο, ε, στην ε, λονδινο Λονδίνο-Μπέρνιχαμ έχουν αυξηθεί κατά 20%. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο Catch ο κύριος Ντόρφον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα απλώς να σας εξιστορήσω μία προσωπική εμπειρία διότι ε, ε, ήμουνα σε ένα τρένο από το, που περνά από τον Μπρένερ προς τη Βερόνα ε, και που αφιερωνόταν επί χρόνια η ε, για εμπορευματικές ε, και ε, επιβατικές μεταφορές και υπάρχουν πέντε δρομολόγια την ημέρα από την Αυστρία χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποιος κατάλογος με τις ώρες αναχωρήσεως. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι δεν είναι δυνατόν γίνονται τα πράγματα πιο περίπλοκα όχι από ένα πολύ ουσιαστικό θέμα αλλά από μικρές λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει κάποια κύρωση και να κοιτάξετε να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλοι και να συμμορφωθούν στις οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φερέιρα, ένα λεπτό. Είναι προφανής ο στόχος του συνολικού πακέτου. Ο αρχικός ε, στόχος ήταν η βάση της, να τεθούν βάσει της διαλειτουργικότητας. Όμως από τότε είχαμε πει ότι στην πραγματικότητα ε, θέλαμε, ο στόχος ήταν να ανοιχθεί ο τομέας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Όπως και άλλες φιλελευθερώσεις, ε, ξεκινάς υπογραμμίζοντας το τι δεν λειτουργεί εκείνη τη στιγμή και καταλήγεις στην διάλυση του δημόσιου τομέα, στο άνοιγμα, σε, στο λεγόμενο ανταγωνισμό και στην πλήρη καταστροφή τελικά. Η απελευθέρωση είναι η, ο, η αιτία και όχι η λύση των προβλημάτων τελικά. Πλήττονται και οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι. Ε, δεν θα διαφωνούσα υπό την προπόθεση ότι θα είχαμε στο μυαλό μα οικολογικού και άλλου παράγοντε. Όχι όμω να παραδώσουμε του σιδηροδρόμου στα ιδιωτικά συμφέροντα μέσω τη απελευθέρωση ε, της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Τι κάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω στην κατάσταση ε, των, ε, των ατόμων ε, που εργάζονται στο σιδηροδρομικό τομέα κατά την περίοδο της κρίσης, διότι στη Ρουμανία είχαμε 6.000 απολύσεις το κοινωνικό ταμείο και το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση θα κινητοποιηθούν για να βοηθήσουν. Θα ήταν όμως καλός να υπάρξει μία στρατηγική μακροπρόθεσμη για την εξέλιξη των σιδηροδρόμων κατά τρόπον ώστε να υπάρξει κατάλληλο προσωπικό και να μπορεί να προστατευτεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπο Κάλλα, για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και την αναθεώρηση του πρώτου πακέτου. Θα ήθελα απλώς τώρα να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, η ενημέρωση για τα 21 κράτη-μέλη και τους συγκεκριμένους λόγους γιατί έχουμε στείλει αυτή την αιτιολογημένη γνώμη, όλα αυτά τα στοιχεία είναι δημόσια. Οποιοςδήποτε μπορεί να ενημερωθεί λοιπόν. Αυτό το πρώτο συνδρομικό πακέτο είχε καλές προθέσεις να καταργηθούν τα εμπόδια και να βελτιωθούν οι συνθήκες για να λειτουργήσουν με καλύτερο τρόπο οι μεταφορές. Τον ίδιο στόχο θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε και με την αναθεώρηση του πακέτου. Το πρόβλημα δεν ήταν κακό το πακέτο, αλλά προβληματική ήταν η εφαρμογή του και ανεπαρκής. Και επομένως ε, παραμένουν τα εμπόδια και οι αντιστάσεις στην κατάργησή τους είναι πολύ μεγάλες. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα ε, με κρατικά μονοπόλια, έλλειψη διαλειτουργικότητας, επομένως πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη διαλειτουργικότητα και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος της μεταρρύθμισης ε, των σιδηροδρόμων. Το πρόβλημα είναι ότι η μεταρρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά θα πρέπει να εξορροπήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια με ποιοτικού ελέγχους. Ε, στο πακέτο ε, έχουμε σκεφτεί πώς θα ενδυναμώσουμε το ρόλο των ρυθμιστικών φορέων. Το πρόβλημα είναι ότι ο ρόλος τους ε, εμπλέκεται με τα συμφέροντα των κρατικών εταιριών, επομένως ο έλεγχος είναι όχι ο ιδανικός. Όλα αυτά τα θέματα θα τα αντιμετωπίσουμε με την αναθεώρηση του πακέτου των σιδηροδρόμων και με κάποια στρατηγικά κείμενα που θα εκδώσουμε και κατάλληλη χρηματοδότηση. Κάτι που είναι ένα μείζον πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε καινοτόμους ε, τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πολλοί βουλευτές ε, μίλησαν για την ανάγκη ξένων επενδύσεων. Πρέπει να συνδυάσουμε όλα τα εργαλεία και να βρούμε και νέα εργαλεία, ούτως ώστε να υπάρξουν νέοι πόροι για επενδύσεις στους σιδηροδρόμους, ε, μοντέρνα συστήματα διαχείρισης, συστήματα κρατήσεων για να αγοράζουμε εισιτήρια με αντίστοιχο τρόπο όπως τα αγοράζουμε στις ε, εναέριες μεταφορές. Καλύτερη σύνδεση επίσης της Ανατολικής Ευρώπης με τη Δυτική Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και αυτό παραμένει ένα πρόβλημα. Θα μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες, θα μπορούσα να μακρηγορήσω. Θα μπορούσα να αναφέρω όλα τα στοιχεία τα οποία είναι σε φάση επανεξέταση στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του πακέτου, αλλά θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις όταν συγκεκριμενοποιηθούν τα νομοθετικά κείμενα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και με την παρέμβασή σας Ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση και επανερχόμαστε στην ε, ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε μια άλλη ε, προφορική ε,